Καλώς Καλώ ήρθατε λοιπόν στην νέα κοινή συνεδρίαση Επιτροπή Προπολογισμών και Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Σήμερα έχουμε μία ε, παρουσίαση του λεκτικού συνεδρίου, γρήγορη ανάλυση τη κατάσταση ε, για τις ε, εκκρεμή αναλήψη υποχρεώσεων στην Ευρώπη των 27. Η κατάσταση είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους. Η συνεδρίαση αναμεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Υπάρχει διερμηνία. Τώρα, τα πρακτικά της 27 Νοεμβρίου και της, 10 και, και της 7 Δεκεμβρίου θα εγκριθούν αν δεν διατυπωθούν ενστάσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Καλωσορίζω το μέλος του ηλεκτρικού συνεδρίου, την κυρία Ιβάνοβα. Η συγητή για το θέμα αυτό είναι ο κύριος Πυρίνσκι. Διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το έγγραφο. Είναι αρκετά δύσκολο ε, στόχος είναι να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών για τις για την δίκαιη κατανομή των πόρων στους ε, φακέλους του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Έχω μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσω την παρουσίασή σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχετε απόλυτο δίκιο ήταν ένα από τα δυσκολότερα έγγραφα τα οποία καταρτήσαμε. Η ίδια η έκθεση δεν είναι τόσο δύσκολη. Πρόκειται για μια ε, ανασκόπηση των ε, εκκρεμωτήτων σχετικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Η διαδικασία λοιπόν ε, έχει αρκετές προκλήσεις. Όταν προσπαθούσαμε να σκεγγραφίσουμε τα κυριότερα βήματα στην ε, κατανομή των ε, τα, πόρων από το Ταμείο Συνοχής. Κοιτάξαμε λοιπόν ε, διάφορες ε, πηγές πληροφοριών έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση της ε, κατανομής των πόρων στα κράτη-μέλη. Θα εστιάσω λοιπόν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιτισμοσομικό πλαίσιο 2021-2027. Η διαδικασία έχει παραμείνει σχεδόν ίδια σε σχέση με το 2006 θα ξεκινήσω λοιπόν αμέσως με την παρουσίασή μου. Για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν προπολογισμό 373 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πολιτική συνοχή, κάτι δηλαδή που, που είναι 10% λιγότερο από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, 2014 με 2020. Όπω και στι προηγούμενε περιόδου, έτσι και εδώ θα δείτε ότι τα κονδύλια θα διοχετευτούν μέσω τριών ταμείων, ERDF, ESF, ε, και Ταμείο Συνοχής. Όπως βλέπετε επίσης από τη διαφάνεια έχει προταθεί 46,7 δισεκατομμύρια ευρώ να ε, ανήκουν στο Ταμείο Συνοχής και στο Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ ε, να διατεθεί το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή 326,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα δύο ταμεία Περιφερικής Ανάπτυξης και Κοινωνικό Ταμείο Πλάς θα ε, σπάσουν σε δύο Τομεί επενδύσεις σε θέση εργασίας και ανάπτυξη και ε, τον στόχο εδαφικής συνεργασίας. Τώρα, πού προκύπτουν οι περιπλοκές με, ε, από τις διαφορετικές ε, διαδικασίες που προκυπτουν οι περιπλοκες απο τις διαφορετικες διαδικασιες που χρησιμοποιουνται για την διάθεση των πόρων. Ας ξεκινήσουμε με την διαδικασία που διέπει την χορήγηση κονδυλίων για επενδύσεις. 85% του συνολικού ε, ποσού που διατίθεται για τη συνοχή. Για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, λοιπόν, ω αφετηρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να συνεχίσει η κατηγοριοποίηση των ε, περιφερειών της Ευρώπης σε τρεις κατηγορίες. Τις λιγότερο αναπτυγμένες, τις ε, περιφέρειες σε μεταβατικό στάδιο και τις αναπτυγμένες. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού υπάρχει ή, υπάρχουν σε ή μεταβατικές όπως το ονομάζονται περιφέρειες. Έχουν εντοπιστεί πέντε τέτοιες περιφέρειες με ε, μέσο όρο ΑΕΠ μεταξύ 75 και 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο στοιχείο λοιπόν είναι ότι για την περίοδο 2021-2027 η πρόταση είναι να διευρυνθεί η κατηγορία αυτή και να συμπεριλαμβάνει όλες τις περιφέρειες με ΑΕΠ μεταξύ 75 και 100% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυξάνεται λοιπόν το 90% γίνεται 100%. Οι περιφέρειες ε, λοιπόν αυτές που προηγουμένως ανήκαν στην κατηγορία περισσότερο ανεπτυγμένε, τώρα άλλαξαν κατηγορία, υποβιβάστηκαν σε μεταβατικές περιφέρειες. Περίπου 10% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, θα επηρεαστεί από αυτές τις αλλαγές. Το αποτέλεσμα και ο αντίκτυπος αυτές τις ε, περιφέρειες σε μεταβατικό στάδιο θα είναι θετικό. Δηλαδή θα λάβουν περισσότερη χρηματοδότηση από τις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες. Επίσης, Χρησιμοποιούνται διαφορετικές διαδικασίες για την διάθεση των πόρων ε, ανάλογα την κατηγορία. Δηλαδή για τις, πιο, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες ακολουθείται μία μέθοδος, για τις ε, μεταβατικές άλλη και αντίστοιχα διαφορετική για τις ε, πιο ανεπτυγμένες. Θα προσπαθήσω λοιπόν με απλά λόγια να σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε μία από αυτές τις περιφέρειες. Αρχίζουμε με τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες όπου ορίζονται ως τέτοιες οι περιφέρειες όπου το ΑΕΠ τους είναι μέχρι το 75% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ βλέπετε ένα πλασματικό κράτος μέλος, δεν υπάρχει αυτό. Βλέπουμε πρώτα ότι γίνεται ένας υπολογισμός του, συνολικού ε, προβλη... χάσματος ευημερίας σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα δεύτερο στάδιο μια συνιστόσα από διάφορες ε, συνισταμένες στην περίπτωση αυτή έχουμε 1,3% του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος, δηλαδή ε, διαφορετικές μετά συνισταμένες που βασίζονται στον σχετικό πλούτο και επιτρέπουν σε μία λιγότερο ή περισσότερο φτωχή χώρα να λάβει διαφορετική χρηματοδότηση. Αυτές οι συνιστώσεις έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με την, περίοδο, με την προηγούμενη περίοδο 2014-2020. Το τρίτο στάδιο που ακολουθεί τα δύο αυτά ποσά είναι τα είναι τα πριμ που χορηγούνται για εκπαιδευτικού στόχου, για καταπολέμηση τη ανεργία. Για την περίοδο 2014-2020 υπήρχε ένα τέτοιο μόνο ποσό για την καταπολέμηση της ανεργίας, ενώ τώρα τα κριτήρια έχουν διαφοροποιηθεί. Για την περίοδο 2021-2027 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δύο τελείως διαφορετικά πριμ, για τη μετανάστευση και την ε, μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για όλα αυτά, αλλά όποιος ε, θέλει έχω στη διάθεσή μου τις ε, πληροφορίες αυτές. Μετά, άλλος τύπος περιφέρειας. Θα πάμε στο αντίθετο άκρο στι πιο αναπτυγμένε περιφέρειες και θα αφήσουμε τι ε, περιφέρειες σε μεταβατικό στάδιο για το τέλο, γιατί είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Για τι πιο αναπτυγμένε περιφέρειες λοιπόν το ε, ε, είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλάζει τελείω το σκεπτικό για την κατανομή των πόρων. Φυσικά εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτή η διαφορά ως προς την ευημερία των πολιτών αλλά έχουμε την χρηματοδότηση στο σύνολό της για όλες τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε ότι οι επιμέρου, μεμονωμένες πιστώσεις βασίζονται στο, στα συνολικά ποσά για 7 διαφορετικούς ε, τομείς. 7 δείκτες δηλαδή που έχουν να κάνουν με την ανεργία, με την ε, ε, εκπαίδευση, με εκείνους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, με το αέπανα περιοχή και την πυκνότητα του πληθυσμού. Όλοι αυτοί οι δείκτες έχουν διαφορετικό βάρος στον υπολογισμό μας. Χρησιμοποιούμε μόνο έναν από αυτούς ε, τους ε, δείκτες, για παράδειγμα, τον πληθυσμό. Εδώ υπάρχει ε, μια στάθμιση του 20, της τάξης του 20% βάσει της οποίας υπολογίζουμε το 100% της χρηματοδότησης βασισμένο σε, στο ποσό των 18 ευρώ ανακεφαλή αυτό το ποσό, τα 18 ευρώ, ε, βρίσκεται στο παράρτημα του κανονισμού περί κοινών διατάξεων. Πολλαπλασιάζουμε λοιπόν με το 7 την επταετή περίοδο και προκύπτουμε στο 26, στα 26 δισεκατομμύρια για όλες τις ε, πολύ αναπτυγμένες περιφέρειες. Δεύτερος υπολογισμός, εκεί όπου το σύνολο του πληθυσμού πολλαπλασιάζεται από τη στάθμιση του ε, δίκτυ, 20% σε αυτήν την περίπτωση. Τώρα, η διαφορά με τις ε, λιγότερο αρνητικμένες περιοχές είναι ότι και εδώ υπάρχουν τα πριμ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Όμως εδώ αφορούν δύο νέους τομείς, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και μετανάστευση. Μπορούν λοιπόν να προσθεθούν αυτοί οι δύο τομείς όπου χρειάζεται σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2014-2020 έχουν γίνει αλλαγές ως προς τη στάθμιση των διαφορετικών δικτών και την ε, προσθήκη των, ε, των καινούριων πριν. Φυσικά υπάρχει το παράρτημα με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες στα έγγραφά σας. Περνάμε τώρα στις μεταβατικές περιφέρειες. Είναι το πιο δύσκολο και περίπλοκο στάδιο της διαδικασίας αυτής, διότι εδώ πρέπει να γίνουν πολύ περισσότεροι υπολογισμοί. Φυσικά βλέπουμε ότι υπάρχουν στοιχεία και από τις ε, προηγούμενες δύο κατηγορίες περιφερειών, τις λιγότερο και περισσότερο αναπτυγμένες. Οπότε έχουμε συνδυάσει την μεθοδολογία για αυτές, από αυτές τις δύο περιφέρειες και έχουμε προσπαθήσει να την παρουσιάσουμε εδώ. Ε, λοιπόν, για, για μια μεταβατική περιφέρεια το σημαντικό είναι να δούμε ότι υπάρχει ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο επίπεδο στήριξης ανακεφαλή. Υπάρχουν κατά ποσά, ελάχιστα ποσά, 18 ευρώ, όπως προβλέπει ο κανονισμός, και το μέγιστο εδώ είναι πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί απαιτεί έναν πιο δύσκολο υπολογισμό και το ποσό αυτό είναι 80 ευρώ κατά άτομο. Αυτό το ποσό όμως δεν είναι κατά αποκοπή, μπορεί να διαφέρει. Και ο υπολογισμός του ποσού αυτού είναι το 60% των κονδυλίων κατά κεφαλή περιφερειών με μέσο όρο ΑΕΠ 75 Έτσι προκύπτουμε στο, στα 80 ευρώ κατά άτομο. Βέβαια, για διαφορετικά ποσοστά ΑΕΠ ενδιαφέρει και το ποσό. Αν συγκρίνουμε τώρα τη διαδικασία αυτή με τη διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, θα δούμε ότι έχουν γίνει αλλαγές στον υπολογισμό του θεωρητικού ανώτατου επίπεδου πιστώσεων. Έχει γίνει μια αύξηση από 40% σε 60% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Η γραμμή που βλέπετε ανάμεσα στο ανώτατο και στο κατώτατο ε, αφορά αυτήν την υποθετική περιοχή. Αντιπαραβάλλεται λοιπόν το ΑΕΠ αυτής της ε, περιφέρειας με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ βλέπουμε ένα, μέσο, ένα επίπεδο 87,8% που αντιστοιχεί στην ε, στήριξη κατά τα άτομο 50 ευρώ. Αυτά τα 50 ευρώ πολλαπλασιάζονται με το σύνολο του πληθυσμού μιας περιφέρειας. Το ξέρω πως σας φαίνονται περίπλοκα όλα αυτά, αλλά θα βρείτε εξήγηση και περισσότερες λεπτομέρειες στο έγγραφό σας. Βλέπω πως ήδη έχω μιλήσει 12 λεπτά και ούτε στα μισά δεν έχω φτάσει της παρουσίασής μου, όμως νομίζω πως αξίζει τον κόπο, αν μου επιτρέψει και η κυρία Πρόεδρος, να σας παρουσιάσω εν συντομία τους υπόλοιπους στόχους, δηλαδή την, ε, το στόχο της εδαφικής συνεργασίας. Όπως βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια, έχουμε υπολογίσει τις πιστώσεις με βάση ποσά που εξαρτώνται από την εδαφική διασυνοριακή συνεργασία, την ε, συνεργασία στη θάλασσα, διεθνική συνεργασία και την συνεργασία μεταξύ των ε, εξόχως απόκεντρων περιοχών. Τα ποσά εδώ είναι αμεληταία σε σχέση με τις προηγούμενες κατηγορίες. Είναι μόλις το 2,5% του συνολικού προϋπολογισμού. Τώρα, λίγα λόγια για το Ταμείο Συνοχής. Να σας πω ότι εδώ παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το νέο στοιχείο είναι ότι έχουμε εισαγαγεί ένα ανώτατο όριο για την επόμενη περίοδο. Η συνεισφορά των κρατών μελών θα περιοριστεί στο 1 τρίτο των του συνόλου των, των πιστώσεων που λαμβάνουν. Τουλάχιστον το 1 τρίτο λοιπόν πήγαινε στο Ταμείο Συνοχής, τώρα είναι το ανώτατο όριο αυτό το 1 τρίτο. Τώρα, στις αρχικές πιστώσεις γίνονται και τροποποιήσεις. Έχει οριστεί το ανώτατο όριο που μπορεί να λάβει ένα κράτος μέλος και το ελάχιστο όριο. Αυτά λοιπόν είναι τα ε, όρια, καθώς επίσης και ένα δίχτυ ασφαλείας που υπάρχει. Τώρα, αν έχετε ερωτήσεις, θα σας απαντήσω σχετικά με αυτό αργότερα. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε την εξέλιξη των πιστώσεων ανάλογα με τον τύπο της περιφέρειας. Συγκρίνουμε την προηγούμενη με την ε, επόμενη περίοδο προγραμματισμού και βλέπουμε τη μείωση στο Ταμείο Συνοχής, όπου συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μεν μείωση αλλά αντισταθμίζεται από τις αλλαγές που έχουν γίνει στο ε, Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης και το Κοινωνικό Ταμείο σε συνδυασμό με τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Εκεί στις ε, έχει παρατηρηθεί αύξηση και ε, παρά το ότι έχω ακόμα κάποια σχόλια να κάνω, εν είδη συμπεράσματος, θα σταματήσω εδώ για να ε, μην ξεπεράσω το χρονογόρευση και να σας πω ότι με τα χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι το έγγραφο αυτό είναι σαν ε, λευκή σημαία είναι πάρα πολύ σημαντικό, το διάβασα με προσοχή και θεωρώ πως είναι σημαντικό διότι δείχνει ότι η ε, κατανομή των πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να γίνει πιο δίκαιη. Το σκεπτικό του επόμενου πολιετού σε δημοσιονομικού πλαισίου έχει αλλάξει σε σχέση με το προηγούμενο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ισότητα ως προς την αντιμετώπιση των ε, κρατών μελών και κάθε αλλαγή έχουμε παρατηρήσει, έχουμε διαπιστώσει ότι οδηγεί σε ανισότητες. Ο κύριος Πυρίνσκι που είναι ο εισηγητή, θα λάβει τώρα το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστώ και την κυρία Ιβανό. Μια πολύ γενναία προσπάθεια. Και την προσπάθεια μέσα σε 15 λεπτά να μας κάνει επισκόπηση ενός άκρος πολύπλοκου, όπως είπε και η ίδια, όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε. φυσικά πρέπει να έχουμε υπόψη όταν συζητούμε αυτή την αναθεώρηση το γενικό ζήτημα της δικαιοσύνης. Το είπατε και εσείς. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και το τελευταίο και προηγουμένως για τα ταμεία συνοχής και τη διάθεση των κονδυλίων αυτών με δίκαιο τρόπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το στόχο της αξιολόγησης αυτής και να αντιληφθούμε με ποια διαδικασία καθορίζονται τα ποσά που είναι διαθέσιμα για τα κράτη-μέλη. Τη συλλογιστική δηλαδή της όλης διαδικασίας, αλλά και τη συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή. Που οδηγεί δηλαδή στην πράξη αυτή συλλογιστική. Υπάρχει ένα τμήμα που έχει να κάνει με την επισκόπηση της διαδικασίας. Ε, το καλύψατε 3,73 δις ευρώ ε, είναι το πόσο που διατίθεται 10% λιγότερο εν παρόδο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και υπάρχει αυτή η διαίρεση έκτα και ε, ετπα από τη μία και συνοχή από την άλλη. Σε αυτή την επισκόπηση αναφέρεται ότι ο στόχος του εγχειρήματο είναι η οικονομική, κοινωνική και δαφική συνοχή. Στην πράξη και σε σχέση με την προκειμένη έκθεση αυτό σημαίνει να μειωθεί το χάσμα ευμερίας ως προς την ευημερία. Δηλαδή. Και αν θυμηθεί κανείς και τα τέσσερα κριτήρια τα οποία χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ένα έχει ακριβώς να κάνει με την ευημερία, γιατί είναι ο σχετικός πλούτος, Δεύτερο είναι ανεργία, εργασία, εκπαίδευση, δημογραφικά κριτήρια ή όλοι αυτοί δέσμοι και δύο νέα. Κλίμα, πράσινες εκπομπές ε, και μεταναστευτικές ροές στο τέταρτο. Και το πρώτο ερώτημα που προκύπτει εδώ, κυρία Πρόεδρε, είναι πώς και έτσι. Γιατί αυτά τα δύο νέα κριτήρια έχουν άμεση σχέση με τη συνοχή ή μήπω πρόκειται για ζητήματα που θα έπρεπε να τα είχαμε αντιμετωπίσει διαφορετικά και όχι εγγράφοντας τα στον προβλήμα της συνοχής. Κύριε Βανόβα τώρα μας περιέγραψε τη διαδικασία της ανάθεσης. Θέλω να σας υπενθυμίσω τις τρεις βασικές ε, στάσεις, ε, μάλλον τα τρία βασικά στάδια, η αρχική, ανάθεση, προσαρμογές και μια τρίτη, ένα τρίτο στάδιο που αναφέρεται είναι το παζάρεμα, αν θέλετε, διαπραγμάτευση όπου εκεί πλέον βγαίνουμε από τα κριτήρια και μπαίνουμε στην πολιτική διαπραγμάτευση, το παζάρεμα που είναι και τελική φάση. Δεν είναι το αντικείμενο αυτή τη εξόλεξη, αλλά αναφέρεται. Σε ό,τι αφορά την αρχική ανάθεση κατανομή, είπε πολύ καλά κύριε Βανόβα νομίζω, ποιοι είναι οι δύο στόχοι σε ό,τι αφορά καταρχάς ανάπτυξη και απασχόληση και την εδαφική συνεργασία. Βέβαια, εργασία και ανάπτυξη είναι ο βασικός στόχος. 316,8 δις. και το βασικό κριτήριο είναι ο σχετικός πλούτος. Υπολογισμό ε, του κατακεφαλήνα να έπια μια δεδομένη περιφέρεια απέναντι σε σχέση με το μέσο όρο στην Ένωση και τρεις κατηγορίες περιφερειών. Μας τα πει κυρία Ιβανό. Εδώ νομίζω κυρία Πρόεδρε πρέπει να αναφέρουμε το δεύτερο στάδιο που είναι τρία για τις λιγότερο επιτυγμένες που είναι ο συντελεστής που εφαρμόζεται τα είπε η κυρία Ιβανόβα δεν εξαρτάται από το ΑΕΠ αλλά από το εθνικό καθάριστο εισόδημα αυτός ο συντελεστής για αυτοί οι συντελεστές τέλο πάντων μερίδιο του ε, εισοδήματος 82 99 πάνω από 82 το πάντων τεχνικό στοιχείο αλλά έχει σημαντικές επιπτώσεις και τελικό ποσό το τελικό ποσό επηρεάζεται για τις ε, περιφέρειες που βρίσκονται σε φάση μετάβασης μας τα είπε πάλι κύριε Βανόβου πολύ ξεκάθαρα. Το μόνο που θέλω εγώ να προσθέσω, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι αυτή η επέκταση 10% στο 100% τελικά τη Γαλλία, τη Φιλανδία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία και την Ολλανδία οφείλει. που αντιμετωπίζονται ω μεταβατικές και όχι ανεπτυγμένε οι περιφέρειες. Και έχουμε βέβαια και τα τρία αυτά στάδια της πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Μας τα είπε η κυρία Ιβανόβα. Το εδαφικό κριτήριο εδώ και ο πληθυσμός είναι το σημαντικό και έχουμε και του επτά δείκτες που προσαρμόζουν αρχέ εκτιμήσεις ε, εδαφική συνεργασία, 9,5 δις ε, από το ΕΤΠΑ, 4 σκέλη, εξάρτητα τον πληθυσμό. Η συνοχή, κυρία Πρόεδρε, η συνοχή μεταξύ των κρατών καλύπτεται βέβαια από τα ταμείο όπως το είπε και η κυρία Ευανόβα. Εδώ βλέπουμε μεγάλη μείωση 46,7 δις το ποσό για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού και επιλέξιμα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία το καθάριστο εθνικό εισόδημα είναι ε, μέχρι το 90% του μέσου όρου της Ένωσης. Ε, υπάρχουν τέσσερα βήματα για να φτάσουμε στην ανάθεση, του, στην κατανομή των κονδυλίων. Ένα υπολογισμό του συνολικού ποσού με βάση 62,90 ευρώ κατά κεφαλή και το πολλαπλασιάζουμε το πληθυσμό πεμπίτη στο πεδίο. Αυτό. Να συντομεύετε κύριε Πίνης, κύριε Πρόεδρος. Ναι. Θα σταματήσω τότε εδώ και θα ρωτήσω τα 5-6 ερωτήματα που είχα να θέσω στην Κομισιόν. Το πρώτο ερώτημα. Γιατί από το 92% στο 100% σε ό,τι αφορά την κάλυψη για τις περιοχές που βρίσκονται στη φάση μετάβασης. Γιατί έτσι όπως τα λέτε στην έκθεση υπήρχε φαίνεται μια ανησυχία σε ό,τι αφορά λιγότερο ανεπτυγμένες και την απόσταση από τις πιο ανεπτυγμένες. Δεν είναι και τόσο καλή αυτή η εξήγηση κατά την άποψή μου. Γιατί υπάρχει μείωση για μείζονε επενδύσει και για τι υποδομέ των μεταφορών, κάτι αναγκαίο στο τομέα, λέτε, τη συνοχή. Και δίνεται μια εξήγηση για τα 13 νέα κράτη που δεν λέτε χρειάζονται τόσε ε, επενδύσεις ο περιβάλλον και υποδομές. Μα αν κοιτάξει κανείς τα διευρωπαϊκά δίκτυα, δίκτυα, θα δει, κυρία Πρόεδρε, ότι υπάρχει απόλυτη ανισορροπία σε ό,τι αφορά την πυκνότητα του δικτύου μεταξύ Κεντροανατολική Ευρώπη και Δυτική Ευρώπη. Άρα καθόλου καλή η εξήγηση για τη μείωση 45% εδώ. Τρίο και, το, και τέταρτο κριτήρια. Κλίμα και μετανάστευση το είπα και ρωτώ γιατί. Γιατί έχουν ενσωματωθεί στην πολιτική συνοχή. και όχι σε μια άλλη. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα ετοιμότητα των κρατών μελών. να απορροφήσουν επιτυχώς τα ποσά δεδομένης της ανάγκης συγχρηματοδότησης και διαχείρισης. Και βεβαίως κύριε Πρόεδρε υπάρχει και το συνολικότερο θέμα των δεδομένων. Υπάρχει ένας χάρτης στην αναθεώρηση αυτή που μας δείχνει τι γίνεται με την ταξινόμηση των περιφέρειων για την επόμενη ε, περίοδο και χρησιμοποιούνται στοιχεία του 2016. Πώς έχει κατάσταση. Ερωτηματικό. Και το τελευταίο ερώτημα. Κάτι που αναφέρατε νομίζω και εσείς κυρία Πρόεδρε για πρώτη φορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε και τη μεθοδολογία. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε διότι είναι ένα τεράστιο βήμα προς διαφάνεια. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Ο Ντέρεκ Βον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο που ήθελα να πω απόψε ελέγχου τον προπολογισμό ότι είναι καλύτερα να κοιτάμε προς τα μπροστά αντί για προς τα πίσω. Αυτό πρέπει να κάνουμε τον προπολογισμό. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Ιβανόβα για την παρουσίαση αυτού του περίπλοκου ζητήματος. Είναι περίπλοκο και αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Αυτά τα νέα κριτήρια που ανέφερε ο κ. Πυρίνσκι, ειδικότερα για την κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση, ίσως θα πρέπει να αποτυπώνονται κάπου στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, διότι είναι νέα ζητήματα. Πιστεύω ότι ίσως να περιπλέκουμε περισσότερο ακόμα τώρα τη κονδέλια. Ίσως πρέπει να τα κάνουμε πιο απλά, να είναι ευκολότερο να τα καταλάβει κανείς και να εξηγούμε γιατί υποστηρίζουμε αυτά τα νέα δύο ζητήματα. Δεν ξέρω αν το λεκτικό συνέδριο συμφωνεί μαζί μου ότι αυτά τα περίπλοκα πράγματα πρέπει να τα προσθέσουμε Το δεύτερο το συνολικό κονδύλιο για την πολιτική συνοχή. Προφανώς υπάρχει μείωση και εδώ ζητώ συγγνώμη για άλλη μια φορά για το Brexit, διότι όπως φαίνεται αυτό επηρεάζει το μελλοντικό ΠΔΠ. Βλέπουμε κάποιε περικοπές που προτείνονται για κράτη-μέλη, διότι το... δημιουργήθηκε ουσιαστικά περικοπή σχεδόν 24% για ορισμένα κράτη-μέλη, που είναι τεράστια Πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτέ οι περικοπέ έγιναν στο σωστό επίπεδο, γιατί όπω είπαμε είναι τεράστιε περικοπέ 24%. Και το τελευταίο που είχα να πω αφορά αυτό που είπε ο κύριο Πυρίνσκι ε, για το πρόγραμμα. Έχουν γίνει πολιτικέ συζητήσει μέχρι το τέλο των διαπραγματεύσεων. Την προηγούμενη φορά, συνάδελφοι, έτρεχαν ε, τελευταία στιγμή. Θυμάμαι στην τελευταία τελευταία σύνοδο κορυφή ε, για τι διαπραγματεύσει του παρόντο ΠΔΠ και διάφορα κράτη-μέλη λαμβάνουν εκατομμύρια ε, ε, ε, επιπλέον χωρί καμία μέθοδο, χωρί καμία διαφάνεια για την ΚΑΠ, για άλλα θέματα. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Ξανά, αυτό θα πρέπει να εξετάζει η Επιτροπή Έλεγχου του Προπολογισμού. Αλλά και το ελληνικό Συνέδριο θα πρέπει να ε, ε, επαγρυπνεί ώστε να έχουμε ένα διαφανέ ΠΔΠ στο τέλο τη διαπραγματευτική διαδικασία, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα κράτη-μέλη θα υποστηρίξουν το ΠΔΠ. Uh-huh. Μαλετίτς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία ε, Ιβανόβα για την άριστη παρουσίαση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό τον προτινόμενο συντελεστή όσον αφορά την εθνική ευημερία, διότι βλέπουμε ότι παρατηρείται μείωση της εθνικής ευημερίας, του συντελεστή αυτού εθνικής ευημερίας και ωραία το σύνολο το συνολικό ποσό μειώνεται λόγω του ότι η Κομισιόν πρότεινε μείωση του συντελεστή. Είναι αυτή η καλύτερη προσέγγιση. Είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος. Αυτός ο νέος τύπος πραγματικά μας επιτρέπει να επιτύχουμε του στόχους, δηλαδή την υποστήριξη των λιγότερων αναπτυγμένων περιοχών. Ειδικότερα όταν βλέπει κανείς το πρώτο κομμάτι του τύπου Ε, για τα επιμέρους απόλυτα ποσά και μετά έχουμε το περιφερειακό πληθυσμό, τον ε, πληθυσμό μιας περιφέρειας ως ε, σημαντικό στοιχείο, έχοντας υπόψη τις δημογραφικές προκλήσεις, τις δημογραφικές προκλήσεις και το γεγονός ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε πολύ ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες χάνουν κόσμο ο οποίος μεταναστεύει σε πιο ανεπτυγμένες χώρες έχουμε λάβει υπόψη στους υπολογισμούς ε, του νέου τύπου όλα αυτά τα στοιχεία. Και μετά τελώς δεν ξέρω αν αυτό το τελευταίο αποτελέσμα τελικά, το τελικό αποτέλεσμα ε, ε, είναι αποτέλεσμα ίσης εφαρμογής όλων των μερών του τύπου σε όλα τα κράτη-μέλη και αν όλοι χρήζουν, έχουν τελικά ίση αντιμετώπιση, μήπως είναι ευνοϊκή αντιμετώπιση για ορισμένους περισσότερο από άλλους. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, παρακαλώ απαντήστε όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου για τι ερωτήσει του. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεση αυτή. Πιστεύουμε ότι μα βοηθά ιδιαίτερα. Εξηγεί καθαρά πώς ε, λειτουργεί η μέθοδος κατανομής. Ελπίζουμε ότι αυτή η παρουσίαση θα βοηθήσει και τις διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, διότι όπως ελπίζουμε τώρα όλοι καταλαβαίνουν τι πρότεινε τουλάχιστον οι Κομισιόν. Από τη δική μας άποψη, η πρόταση είναι σαφής και διαφανής. Ε, το αναφέρατε και εσείς κυρία Πρόεδρε και αναφέρατε και κάποια στοιχεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Επιτροπή πρότεινε έναν προπολογισμό 10% χαμηλότερο για την περίοδο μετά το 2020 από ότι ο σημερινό προπολογισμό. Ε, Γεγονό που σημαίνει ότι προφανώ ε, χρειάστηκαν κάποιε περικοπέ. Δεδομένων αυτών, αν ε, παρατηρήσετε τι προσπαθούμε να επιτύχουμε, πιστεύω ότι τα καταφέραμε πρώτα απ' όλα να δρομολογήσουμε χρήματα περισσότερο σε φτωχέ περιοχέ και κράτη-μέλη. Γιατί θα δείτε από την εκθέση τα τρία τέταρτα του συνολικού ε, προπολογισμού συνοχή πάνε στι φτωχότερε περιοχέ και τα φτωχότερα κράτη-μέλη. Εκεί πρέπει να πηγαίνουν και οι πόροι, μάλιστα, ε, σύμφωνα με την πρότασή μα. Και εκεί πάνε. Επίση, προσπαθήσαμε, αυτό ήταν ο δεύτερο στόχο, ε, να έχουμε μια δίκαιη και ισορροπή κατανομή μεταξύ των κρατών μελών που να αντικατοπτρίζει το επίπεδο ανάπτυξή τους. Ε, αν ε, κάνετε τις αναγκαίες συγκρίσεις θα δείτε ότι υπάρχει κάποια ίση αντιμετώπιση των κρατών μελών ανάλογα με το επίπεδο ευημερία ε, και απασχόληση που επικρατεί εκεί. Και τέλο, για να απαντήσω κάποιε ερωτήσει σα, προσπαθήσαμε να μετριάσουμε και τι ζημίε. Διότι πράγματι σε κάποια κράτη-μέλη, τι απώλειε, συγγνώμη, προσπαθήσαμε να τι σταθμίσουμε. Κάποια κράτη-μέλη θα λάβουν λιγότερα χρήματα από ό,τι λαμβάνουν τώρα. Ο λόγο είναι πολύ απλό αναπτύχθηκαν οικονομικά πολύ θετικά αυτά τα κράτη-μέλη παρά την οικονομική κρίση, το οποίο σημαίνει προφανώς ότι λαμβάνουν λιγότερη στήριξη και θα λαμβάνουν λιγότερη στήριξη στο μέλλον σε σχέση με το, αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεδομένων αυτών, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι το δίχτυ ασφαλεία μα ε, θεωρούμε ότι είναι αρκετά γενναιόδωρο, διότι μιλάμε για μείον 24% σε σχέση με τη σημερινή κατανομή ω μέγιστη ε, αυτή είναι η μέγιστη περικοπή. Είναι πράγματι σημαντική, είναι υψηλή, αλλά ε, για το 2014-2020 είχαμε ε, σχεδόν 45% δίχτυ ασφαλεία. Οπότε κάποια κρατημέλη έχασαν περισσότερο από το μισό δίχτυ ασφαλεία του. Τέλο πάντων, το δίχτυ ασφαλεία μα τώρα είναι πιο γενναιόδωρο από ό,τι έχουμε αυτή, σε αυτή την περίοδο. Ναι, για να απαντήσω κάποιες από τις ερωτήσεις που έθεσαν ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου, γιατί μείωση στο Ταμείο Συνοχής ε, αναφέρθηκε από τον εισηγητή, από την εισηγήτρια κάποιοι λόγοι που το προτείναμε. Θα επενδύσουμε πρώτα απ' όλα σε υποδομές μεταφορών με το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης. Από το 2007 μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου πάνω από ένα δισεκατομμύριο σε υποδομές μεταφορών. Και να ξέρετε ότι έχουμε ένα νέο μηχανισμό τώρα διαθέσιμο, το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη, και πιστεύουμε ότι για την πολιτική συνοχή στο μέλλον θα πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στην καινοτομία στις δεξιότητες και λιγότερο στις υποδομές μεταφορών όπως κάναμε μέχρι σήμερα. Δεδομένων αυτών, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάψουμε να χρηματοδοτούμε στο μέλλον τι υποδομή μεταφορών καθόλου μάλιστα. Απλά θέλουμε να αλλάξουμε του σημείο Τώρα για τους νέους ε, ε, δείκτε ε, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και μετανάστευση. Να υπενθυμίσω ότι η στάθμιση είναι πολύ μικρή, 4%. Οι δύο δείκτε δηλαδή μαζί αντιστοιχούν στο 4% του συνολικού ας κοκτέιλ δικτών οι περισσότερες ε, κατανομές βασίζονται σε ΑΕΠ, ε, όπως είπαμε δεν αλλάζει τίποτα εκεί. Τώρα, δεδομένων αυτών, γιατί συμπεριλάβουμε αυτού του νέου δείκτες, διότι πρώτα απ' όλα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο μέλλον η ένταξη των μεταναστών θα αποτελεί μια νέα προτεραιότητα που δεν χρηματοδοτείται στο παρελθόν και αυτή η νέα προτεραιότητα αντικατοπτρίζεται σε αυτό το νέο κριτήριο στον αριθμό δηλαδή μεταναστών που έχουν εισελθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, όπου θέλουμε να υποστηρίξουμε μια σαφή ενεργειακή μετάβαση ε, υπό τη μορφή μιας, ε, ε, οικονομίας μια οικονομία χαμηλών ανθρωπούχων εκπομπών. Μια νέα πρόκληση και για τα δύο ταμεία μα. Θέλουμε λοιπόν αυτό να αποτυπώνεται με λιγότερο, με περισσότερο έντονο τρόπο μια-δυο προσθήκες ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Έχοντας λάβει υπόψη τις διοικητικές δυνατότητες ε, των κρατών μελών για απορρόφηση των κονδυλίων, ναι, το έχουμε λάβει υπόψη. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στη μέθοδο κατανομή μας, κατανομής μας ε, στο πλαίσιο του capping ε, των ανώτατων επιπέδων έχει μειωθεί αυτό από το σημερινό 2,5% σε κάτι μεταξύ του 2,3% και 1,5%. Αυτό αντικατοπτρίζεται εδώ. Δεδομένων αυτών, θεωρούμε ότι στόχος μας ε, είναι να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίε στην απορρόφηση των κονδυλίων. Δεν θέλουμε λοιπόν να περικόψουμε τα κονδύλια, διότι δεν απορροφήθηκαν τόσο καλά ε, λόγω ε, λήψεων στις διοικητικές ικανότητες. Και επίσης μία τελευταία ερώτηση ε, να απαντήσω. Ναι, χρησιμοποιήσαμε τους μεσόρους του 2014-2016. Έχουμε τώρα ε, το 2017 του δείκτες που δημοσιοποιήθηκαν από τη Eurostat, αλλά η Κομισιόν δεν έχει ακόμα λάβει την απόφαση κατά πόσο θα επικαιροποιήσει την πρόταση για το ΠΔΠ ή όχι. Δεν μπορώ να σα πω λοιπόν αυτή τη στιγμή αν θα επικαιροποιήσουμε ή όχι την πρότασή μας. Θα πρέπει αυτό να αποτελέσει το αντικείμενο μια ευρύτερη συζήτηση πέρα τη πολιτική συνοχή, γιατί επηρεάζει ολόκληρο τον ευρωπαϊκό υπολογισμό και όχι μόνο την περιφερειακή πολιτική. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Yeah, vielen ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ιβάνοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλου ε, του αξιωτικού ευρωβουλευτέ για τι ερωτήσει και τα σχόλια. Να σα υπενθυμίσω βέβαια ότι πρόκειται για μία ταχεία ανασκόπηση τη ε, κατάσταση. Είχαμε δυόμιση μήνε χρόνο για να συντάξουμε την έκθεση αυτή. Πολύ σύντομο λοιπόν χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, είμαστε όσο πλήρης θα θέλαμε. Ε, υπάρχει και ένα αρνητικό από όλα αυτά ότι στην έκθεση αυτή δεν υπάρχουν συστάσεις και συμπεράσματα, όπως σε μια κλασική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Οπότε νομίζω πως δεν θα μπορέσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σχετικά με τις εκτιμήσεις μας. Τα στοιχεία είναι δημόσια. Τα συλλέξαμε από πηγές που είναι προσβάσιμες σε όλους και προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό και να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα με τρόπο, φιλικό προς το χρήστη. Τώρα, ένα γενικότερο συμπέρασμα προσωπικό, μια προσωπική εκτίμηση που θα μπορούσα να κάνω, έχει ως εξή. Η διαδικασία είναι σίγουρα περίπλοκη. Και όπως είπε και ο εισηγητής, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τέτοιες πληροφορίες στο πλαίσιο του κανονισμού περί διατάξεων. Το θεωρώ ένα καλό βήμα προς περισσότερη διαφάνεια για τους ε, ενδιαφέρουμενους φορείς, για ε, όσους ε, λαμβάνουν αποφάσεις, για τους πολίτες. Παραμένει βέβαια πολύ δύσκολο και περίπλοκο το ζήτημα, διότι έχουν εισαχθεί νέα κριτήρια, ο τρόπος υπολογισμού έχει γίνει ακόμα πιο περίπλοκος και αυτό αποτελεί και πρόκληση για μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε μέσα 15 λεπτά όλο αυτό. Ίσως θα μπορούσα να απαντήσω στην κυρία Μάλετιτς, η οποία ρώτησε για τις ε, συνιστώσεις, για, για, για τους συντελεστές. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να εξετάζεται από την σκοπιά ενός μόνο δίκτυ, ενός μόνο κριτηρίου. Ο υπολογισμός αυτός λαμβάνει υπόψη πάρα πολλές συνιστώσεις. Και βλέπουμε ότι τα κριτήρια δεν είναι τα ίδια. Εκεί που υπάρχουν αυξήσει όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, στα δίκτυα ασφαλείας, υπάρχει μείωση αλλού. Αυτή η μείωση βέβαια στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές είναι η μικρότερη από τις τρεις. Είναι δύσκολο λοιπόν να υπολογίσουμε από τώρα ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα για όλες τις περιφέρειες. Βέβαια, ναι, σίγουρα υπάρχει, ο στόχο, υπάρχει μείωση του 10%, όμως νομίζω πως δεν είναι τόσο σημαντικό στοιχείο αυτό. Τώρα, σε ό,τι φορά τις πολιτικές διαπραγματεύσεις, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Ο κύριος Βον είπε ότι αυτό εξάλλου δεν αποτελεί κομμάτι της ε, ανασκόπησής μας οι αρχικές πιστώσεις και οι τροποποίησει ήταν το αντικείμενο της ε, μελέτη, Όσοι βέβαια ενδιαφέρονται μπορούν να δουν τη σελίδα 19 του εγγράφου, το παράρτημα 7 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων για την περίοδο 2014-2020. Εκεί αναφέρονται αυτές οι πρόσθετες πιστώσεις για τις οποίες συμφώνησαν τα κρατημέλη. Σε αυτό το στάδιο όμως, ακριβώς επειδή η διαδικασία βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες πέρα από όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Ευχαριστώ. Ναι, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μετά τον Brexit. Αβέβαια τα πράγματα. Προπού, προτού δώσω το λόγο στον κύριο Πυρίνσκι, να καλωσορίσω την κυρία Κάντενμπαχ. Επέστρεψε αφού είχε σπάσει το πόδι τη, ε, συντομότερα από όσο περιμέναμε. Καλώ ήρθατε λοιπόν και κύριε Πυρίνσκι, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως και θέλω να ευχαριστήσω και τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ρέτζη. Ο κ. Βόν νομίζω έθεσε και κάποια ζητήματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω, αλλά θα ήθελα να εστιάσω στο χάσμα ε, ευημερία, αυτή την έννοια του prosperity gap. Και πρέπει να σας πω κυρία Πρόεδρε ότι και εγώ ε, διαρωτώ με, αν δει κανεί τη σελίδα 15 και το πρώτο παράδειγμα για μια φανταστική περιοχή όπου το χάσμα είναι 10.000 ευρώ μεταξύ δηλαδή του οδήματο ενός ατόμου και του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πληθυσμό 3,5 εκατομμύρια το θεωρητικό ποσό για να κλείσει αυτό το χάσμα είναι 245 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Τελική κατανομή, το τελικό κονδύλιο με τους συντελεστές και τα λοιπά και τα πριν φτάνει στα 3 ε, δύο 2,16 εκατομμύρια. Ξέρω ότι υπάρχει αυτό το κενό που πρέπει να καλυφθεί, 245 δις. Αλλά το ερώτημα της κυρίας Μάλιτιτς, τελικά, μετά από όλο αυτό, την όλη άσκηση και τους υπολογισμού, ο στόχος της συνοχής, δηλαδή η μείωση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών, επιτυγχάνεται. Και νομίζω εδώ ότι στα μελλοντικά βήματά μας θα πρέπει να δούμε πώς αλληλεπιδρά με το InvestEU η συνοχή. Πώς ενσωματών όλα τα εργαλεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας ε, στη νέα περίοδο. Το ελεγκτικό συνέδριο καλά θα κάνει νομίζω να ελέγξει και καλά κάνει και το ελέγχει πώς δηλαδή ε, προχωρά αυτή η όλη διαδικασία και ο χάρτης που θα κοιτάμε στο τέλος της περίοδος ποιο, πού θα είναι η διαχωριστική γραμμή ε, μεταξύ Ανατολής και Δύσης και αν θα είναι τόσο έντονη η διαχωριστική αυτή γραμμή, γιατί τώρα πραγματικά υπάρχει ένας πλήρης διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δύο περιοχών. Πρώτα ευχαριστώ και να μην ξεχνάμε ότι σε 20 ε, χρόνια έχουν μειωθεί κατά το ίμιση οι διαφορές, το χάσμα αυτό Δηλαδή θα ήταν λάθος να δίνουμε υποσχέσεις ότι τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ γρήγορα, όμως ό,τι αφορά τη μεθοδολογία, ε, τουλάχιστον η εξασφάλιση ότι θα προχωρήσουν με δίκιο τρόπο είναι κάτι θετικό. Τώρα, εμείς δεν θέλουμε τώρα να ε, αρχίσουμε τη συζήτηση για όλα τα ταμεία, οι των κρατών και κυβερνήσεων έχουν σίγουρα μπροστά τους ε, ένα δύσκολο χρέος. Θα ευχαριστήσω και το ελεγκτικό συνέδριο και την να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που είναι μια γρήγορη ανάλυση των υπολείπων προς ε, καθάριση και των δυνατοτήτων ε, των κρατών μελών ε, να εφαρμόσουν, να αξιοποιήσουν τα κονδύλια που έχουν στη διάθεσή του. Ο κύριο Σαλαφάκα είναι ο μέρο μα και ο συζητητή και έχουμε δυο κύριο μπομ. Uh, σε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να σας παρουσιάσω αυτή τη γρήγορη επισκόπηση σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα προς εκαθάριση, δηλαδή για τις ε, πιστώσεις που δεν έχουν αξιοποιηθεί, στοιχεία που έχουμε ως το τέλος του 2017. Και έχουμε δημοσιοποιήσει ετήσιες εκθέσεις, ειδικέ εκθέσεις ως ελεγκτικό συνέδριο ήδη ε, τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε υπόψη. Επίσης έχουμε ε, μελετήσει και έγγραφα της Κομισιόν και άλλων οργανισμών. Συναντηθήκαμε πολλές φορές και με την ε, Κομισιόν ε, για να καταλήξουμε αυτό το κτίν. Τα ράλ, τα υπόλοιπα προς εκμετάλλευση είναι δεσμεύσεις, πιστώσεις οι οποίες δεν έχουν ε, αξιοποιηθεί και οι περισσότερες έχουν να κάνουν με κάποια οικονομική υποχρέωση που πρέπει να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό. Ουσιαστικά μεταξύ της έναρξης και της λήξης υπάρχει ένα χάσμα, υπάρχει ε, ένα χρονικό περιθώριο. Πολλές φορές όμως πρέπει να αρχίσουν τα έργα, περνάνε ολόκληρα χρόνια. Και αυτές οι πιστώσεις μπορεί να παραμείνουν σε κρεμότητα για πολλά χρόνια όσο εφαρμόζονται τα project, τα έργα. Σε αυτή την περίοδο θεωρούνται ως υπόλοιπα προς εκαθάριση που αυξάνονται με τις πληρωμές και μειώνονται με τις ε, μάλλον αυξάνονται με τι αναλήψει υποχρεώσεων και μειώνονται με τι πληρωμέ και τι αποδεσμεύσει. Ουσιαστικά μα παρέχει ανάλυση ε, το έγγραφο αυτό για να δούμε τι ε, πρόβλημα υπάρχει και πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Can Όπως μπορείτε να δείτε, μάλλον, όπως μπορείτε να δείτε, Βλέπετε πώς εξελίσσονται τα υπόλοιπα προς εκαθάριση του 2017. Έχουν αυξηθεί από τρεις πτυχές πλευρές σορευτικά έχει αυξηθεί, το βλέπουμε στην γαλάζια γραμμή. Σταδιακά για μια δεκαετία, τα τελευταία χρόνια όμως Έχουμε σημαντική αύξηση. Το 140 που ήταν στα τέλεια του 7 έχει φτάσει σε σχεδόν 270 το 17. 93% αύξηση δηλαδή. Τη μόνη φορά που υπήρξε μείωση ήταν το 2013. Για τεχνικούς λόγους όμως. 20% ήταν το υπόλοιπο προς εγκατάσταση ό,τι αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων το 10, ήταν 25% των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων το 17. Τρίτο στοιχείο, αύξηση των ε, αναλήψεων υποχρεώσεων με διάρκεια πάνω από ένα έτος που αυξήθηκε από 2,1 2,4 μάλλον έτη το 10 σε 2,7 έτη το 2017. Επίσης βλέπουμε σημαντική αύξηση σε τρία επίπεδα. Μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και όπως βλέπετε με την γαλάζια γραμμή, ε, οι κουκίδες, ε, όταν είναι δεκεκομμένη γραμμή δηλαδή, είναι εκτιμήσεις μας μέχρι το 2023. Μετά βλέπετε άνα κατηγορία του 5 βλέπετε για το 17 ότι το 1β ε, τα ήταν το βασικό με 60%. Ο τίτλος 2 14%. Είναι σημαντικό να το βλέπουμε ανακατηγορία, αλλά θα δούμε πώς ε, το ΡΑΛ έχει εξελιχθεί από το 2000 και μετά. Εδώ βλέπετε λοιπόν την εξέλιξη του πολυπροσεκαθάριση αν απειδελταπεί στον κάθε άξονα βλέπουμε το ποσό σε δις ευρώ και στον οριζόντιο άξονα τα έτη χρήσης, τα οικονομικά έτη. Και βλέπουμε ότι υπάρχει αλληλεπικάλυψη σταθερή ε, μια επταετή, στις ε, επταετίες δύο λόγοι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τι αρχέ, στα πρώτα χρόνια ενό δηλαδή πει πολλέ ε, πληρωμέ έχουν να κάνουν με δεσμεύσει που είχαν υποχρεώσει, μάλλον με αναλήψει υποχρεώσεων τη προηγούμενη περίοδου. Επίσης, ε, ισορροπεί η κατάσταση στο τέλος με τις νέες ανάληψεις υποχρεώσεων. Και τα κράτη έχουν περισσότερο χρόνο να, κατα... να απορροφήσουν και να χρησιμοποιήσουν ε, τα κονδύλια. Ενώ είχαν δύο χρόνια πριν, τώρα έχουν τρία. Τώρα, να δούμε τα διαφορετικά και επενδυτικά ταμεία και το σχετικό υπόλοιπο προς εκαθάριση. Βλέπουμε σε επίπεδο κρατών μελών τι ισχύει. Με τα υψηλότερα ραλ έχουμε τρία κράτη που είχαν και υψηλότερες ε, αναλήψεις υποχρεώσεων. Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία. 40% του ραλ το 17 για τα ΕΣΥΦ τα επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία. Και εδώ βλέπετε ότι αν τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν σε σχετικά συγκρίσιμο ρυθμό τα προγράμματα, είναι λογικό το μερίδιο ε, το υπολείπω σε να είναι αναλογικό με το μερίδιο των συνολικών πιστώσεων. Όμω βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίε γιατί υπάρχει απορρόφηση σε διαφορετικού ρυθμού. Και αυτέ τι διαφορέ τι βλέπουμε σε αυτήν τη διαφάνεια για το τρέχον πι. Τα κράτη-μέλη με τα μέλη τα ποσοστά απορρόφηση στα τέλη του 2017 ήταν η Φιλανδία η Αυστρία και η Ιρλανδία, ενώ με το χαμηλότερο ήταν η Ιταλία, Κροατία, η Μάλτα και η Ισπανία. Για να έχουμε λοιπόν μια πλήρη εικόνα του υπόλοιπου σε περιλαμβάνουμε και τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων, τα decommitments. Ανακράτος μέλος και εδώ το βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Ανακράτος μέλος. Λοιπόν, τι αποδεσμεύσεις είχαμε γιατί δεν καταβάλλονται όλες, αποδεσμεύονται για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, αν τα δεσμευμένα ε, ποσά υπερβαίνουν τι συμβατικέ καταληκτικές ημερομηνίε, ή αν το συνολικό ποσό των πληρωμών είναι χαμηλότερο από αυτό το οποίο είχε ε, γραφεί στην σύμβαση. Βλέπετε εδώ, Ρουμανία, Αυστρία, Βουλγαρία έχουν τα περισσότερα ε, ποσοστά, ενώ Πολωνία, Ουγγαρία, Γαλλία έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά. Πρέπει να σα πω ότι το ποσοστό των αποδεσμεύσεων είναι χαμηλό. Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν 2,1% μόλι του συνόλου των ανάληψεων υποχρεώσεων. Τώρα, τι παράγοντες κινδύνους και πιθανές λύσεις έχουμε να αναφέρουμε. Ήδη από το 2002 είχαμε ορίσει κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν το ραλ. Ακόμη και τώρα, το 2019 17 χρόνια μετά ισχύουν τα ίδια. Αλληλεπικάλυψη των 2 πιδελταπή. Πώ επηρεάζει αυτό αυτόματο κανόνα αποδεσμεύσεων και η καθυστερημένη έναρξη των πραγματών. Αυτή είναι οι τρει. Επίση, έχουμε τι απαιτήσει ε, για τα διαρθρωτικά επενδυτικά ε, που έχουν οδηγήσει και σε επίπεδα ρεκόρ ραλ. Με βάση τι εκτιμήσει μα, δε και τι εκτιμήσει κομισιών, το ραλ θα αυξηθεί ακόμη παραπάνω. Οπότε υπάρχει ένας άμεσος κίνδυνος. για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, δεν θα έχουμε επαρκείς πιστώσεις πληρωμών στα τελευταία έτη του ΠΔΠ που ισχύει μέχρι τώρα. Επίση, στην ετήσιε εκθέσει μα ε, λέμε ότι ένα υψηλό ράλ αυξάνει τον κίνδυνο μη φυσιολογικών καθυστερήσεων πληρωμών ανάλογα με αυτό που είδαμε το 2013-2015. Γιατί υπάρχουν ε, πολλέ απαιτήσει πληρωμών που θα αυξηθούν σημαντικά στα τέλη του τρέχοντος ΠΔΠ. Επίσης δεν έχουμε επαρκείς ε, πιστώσεις πληρωμών στο επόμενο ΠΔΠ και έχουμε και μεγαλύτερη έκθεση του προϋπολογισμού της Ένωσης γιατί πέραν των μεκτελεστήσεων, μια απορροφηθησών πιστώσεων έχουμε και το πρόβλημα των νομικών υποχρεώσεων και άλλων liabilities. Ποιες είναι οι λύσεις. Ποιες είναι οι λύσεις. Μπορεί να μειωθεί το υπόλοιπο καθάριση, αν αλλάξει, το πρόσωπο αν αλλάξει το επίπεδο των διαφόρων συνισωσών του προπολογισμού, δηλαδή πιστώσεις, πληρωμών, υποχρεώσεων και αποδεσμεύσει, αν έχουμε αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων που και αν έχουμε χρηματοοικονομική πειθαρχία και πιο απλούς κανόνες για την εκτέλεση του προπολογισμού. Και η βασική πρόκληση βέβαια είναι να μην έχουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο υπόλοιπο προς ε, καθάριση στην τελευταία περίοδο. Δεν έχουμε βρει όμως αυτή τη στιγμή ε, κάποια λύση εμείς. Πρέπει να ληφθούν μέτρα από την Κομισιόν. Εμείς τονίζουμε και στο προηγούμενο έργο μας ποιες είναι οι λύσεις, δηλαδή έγκαιρη έγκριση του νέου ε, ΠΔΠ και των πολιετών προγραμμάτων, απλούστευση των κανόνων, εκτίμηση των αναγκών για πληρωμές και η εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των πιστώσεων πληρωμών και ανάληψη υποχρεώσεων. Αν δεν ακολουθήσει όμως η Κομισιόν τις συστάσεις μας και δεν λάβει μέτρα, θα έχουμε αναπόφευκτα φαινόμενο ως Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοβάμαι πως ε, κινδυνεύουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος με την άλλη φορά. Κύριε Σαλαφράγκα, έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετική αυτή η έκθεση την οποία μας ε, παρουσίασε και εκπώνησε το Ελεκτικό Συνέδριο, γιατί πολύ ξεκάθαρα μας παρουσιάζει τη φύση και τη διάσταση του προβλήματος. Ε, νομίζω το πρόβλημα έχει πώς να το πω, στρατοσφαιρικές διαστάσεις. Είμαστε στις 247 δις και αυτό είναι το 25% των ε, πιστώσεων αλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο των ετήσιων δημοσιονομικών προοπτικών. Είναι πολύ σαφής επίσης η περιγραφή που δίνεται για την προέλευση, για τις αιτίες του προβλήματος. Υπάρχει χάσμα μεταξύ των πιστώσεων ανάπτυξη των και των πιστώσεων πληρωμών, μεγάλη καθυστέρηση εκτέλεση πολλών ε, προγραμμάτων από την Κομισιόν ε, και ε, πληρωμών δηλαδή και επίσης δίνεται και ένα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Υπάρχει μεγάλη επικάλυψη και το λέει και το ελεκτικό συνδέμα μεταξύ των περίοδων εφαρμογής. Επίσης, καθυστερημένη έγκριση των νομοθετικών πλαισίων. Σε ό,τι αφορά την αυτόματη αποδέσμευση ε, και την περίοδο ε, των δύο ετών και που ε, επιμηκύνθηκε. Αν αναλύσουμε τι έγινε το 2002 Είμαστε σε μια περιδίνηση ε, συνεχή, ε, σε έναν κύκλο που επαναλαμβάνεται. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ επιζήμιο για τις λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πολύ σημαντικό νομίζω να λάβουμε υπόψη μας και τους νέους κανόνες ε, του Δημοσιονομικού Κανονισμού του 2018 όπου από την Κομισιόν ζητείται συστηματικά να παράγει προγνώσεις και προγνωστικά και προβλέψεις μακροπρόθεσμες. Δεν θα σχολιάσω αυτές τις απειλές που ανέφερε και το Ελεκτικό Συνέδριο για το προβλέψιμο. Αν υπάρχουν τεράστια υπόλοιπα προς εκαθάριση, θα πρέπει οι καθαρίσεις να γίνονται γέρος, δεν θέλουμε να εκτεθεί ε, οικονομικά η Ένωση υπερβολικά, επομένως μια προτεραιότητα κατά εμά πάρα πολύ σημαντική που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να είναι προφανω η μείωση ε, η δραστική, του υπόλοιπου σε καθάριση. Το ελεγκτικό συνέδριο μας δίνει κάποιες πιθανές λύσεις. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί έχω ξεπεράσει το χρόνο μου. Θέλω όμως να συγχαρώ το ελεγκτικό συνέδριο γιατί πάρα πολύ ξεκάθαρα μας εξηγεί τη σημασία του προβλήματος, τις αιτίε του και τις, τους κινδύνους και τις λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκαρνταθιάμπαλ. Ευχαριστώ πολύ. Είχα στήσει το λόγο γιατί ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με την κατάσταση, με το υπόλοιπο προσεκαθάριση και σε σχέση με τα σχόλια ή τέλο πάντων τις προτάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Το πρώτο, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, είπατε για το 2014, αν κατάλαβα καλά, ότι η μείωση του ΡΑΛ ήταν τεχνικής φύσεως. Ε, διορθώνω, είχα πει το 2013 το 2014 αν αυτό έγινε, έγινε γιατί υπήρξε πολιτική απόφαση ακριβώ. Γιατί είχαμε τον προπολογισμό του 2015 που ήταν μπλοκαρισμένο ακριβώ για να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να βάλουν πιο πολλά χρήματα στι πιστώσει πληρωμών για να καταβληθούν τα 25 δι που εκκρεμούσαν σε απλήρωτου λογαριασμού. Έτσι, για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Επόμενο ναι, πρόεδρο. Ήταν πολύ καλό ο γενικό εισηγητή μα. Ναι, βεβαίω, ο κύριο Ντεπρέ το 2015. Εγώ είχα μπλοκάρει, αλλά το 2014 το κύριο Ντεπρέ που τον βοήθησα έτσι να ξεμπλοκάρει το 2014. Λοιπόν, όπω έλεγα σε σχέση με το ράλι. Από μόνο του το ράλι δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι πολιτικό στόχο. Και το λέω ω προειδοποίηση γιατί κάποιε φορέ με φοβίζει το πώ κάποιοι χρησιμοποιούν το ράλι. Δεν είναι πρόβλημα από μόνο του και καταλαβαίνω το που ο κ. Σαλαφράγκα. Όμως πράγματι θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά ποιε είναι οι αιτίε που οδηγούν σε αύξηση ή μείωση του πολύπου σε καθάριση. Διότι φυσικά υπάρχει χαμηλότερη ταχύτητα εκτέλεση προγράμματο, επηρεάζεται τώρα και αυτό δεν είναι θετικό. Και επομένως υπάρχει Πω δέσμευση και ε, κάποιον δεσμεύσαν μπορώ να το πω έτσι. Άρα το ραλ, το πρόβλημα με το ραλ είναι ότι δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια που είχαν ε, δεσμευθεί. Μα το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι επαρκές οι πληρωμές. Γι' αυτό έχουμε ραλ. Έχουμε λοιπόν αυτή την αναντιστοιχία μεταξύ πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων και σε κάποιες ε, από τις ε, μάλλον σε κάποια από τα συμπεράσματα, ε, πρέπει να πω ότι εκεί δεν συμφωνώ. Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί με τα decommitments, ούτε ξέρω πώς λέγεται στα ισπανικά αυτή η λέξη, ε, και πρέπει να δοθεί γι' αυτό νομίζω πολιτική απάντηση, ενώ το πρόβλημα είναι τεχνικό, άρα αυτό είναι επικίνδυνο. Στόχος είναι οι χώρες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα χρήματα, άρα ο πολιτικός στόχος θα έπρεπε να είναι τα αντικομίτμεντ να μειωθούν ως τον περισσότερο γιατί είναι δράμα με όλο αυτό που μα κοστίζει να βάλουμε κονδύλια στον ευρωπαϊκό περιπολισμό, τελικά να μην μπορούμε για κάποιε περιπτώσει να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια. Και ο, ο μόνο τρόπο από τεχνική πλευρά για να μειωθούν τα υπόλοιπα προσκαθάρισα σε κάποια χρόνια, οι πληρωμέ να υπερβαίνουν τι αναλήψει υποχρεώσεων, δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί Επιπλέον, αν μειώσουμε τι ανάληψει υποχρεώσεων, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Συμβούλιο θα δει ότι υπάρχει μείωση των ανάληψεων υποχρεώσεων και αυτόματα θα μειώσει τι πληρωμέ. Άρα ξαναγυρίζουμε στον ίδιο φαύλο κύκλο. Ο μόνο τρόπο να μειωθεί το υπόλοιπο ψυκαθάριση είναι να αυξηθούν οι πληρωμέ, ώστε σε κάποια χρόνια να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτή τη διαφορά μεταξύ πληρωμών και αναλήψεων υποχρεώσεων. Κύριος Πρόεδρος, κύριε Σαρτουή, ήθελα να χαιρετήσω εγώ τις άριστες αυτές εκθέσεις ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η πρώτη μας επιτρέπει να αποκτήσουμε μια εικόνα των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για την κατανομή των ε, κονδυλίων της πολιτικής συνοχής. Βγήκαμε από τα στεγανά δηλαδή. Ε, πιστεύω ότι θα είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση μεταξύ των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων για να δούμε πώς θα σταματήσουμε ε, το κομμάτι που αντιστοιχεί στον καθένα αυτή την οτροπία. Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε αυτή την κατανομή και δεν θα είναι απλό ούτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις προσπαθώντας να αιτιολογήσει το δίκαιο που αντιστοιχεί στον καθένα αυτό είναι μια αλήθεια αναμφισβητητή. Όσον αφορά τα υπόλοιπα προσεκαθάριση, τα RIL, έχουμε... πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Αν είχαμε υιοθετήσει το ΠΔΠ ήδη τώρα, ώστε όλα να ξεκινήσουν το 2021, δεν ξέρω πώς θα είχαμε αντιμετωπίσει τις πληρωμές. Υπάρχει ε, ένα πρόβλημα ετεροχρονισμού ουσιαστικά. Σας το είχα πει και ε, το έχω ξαναπεί κάποτε ε, κάθε ε, χώρα έχει το δικό του ε, κομμάτι να κάνει όσον αφορά τα περιφερειακά κονδύλια. Εγώ κάποτε ασχολούμουν με τα κοινωνικά χρήματα και μου είπε τότε ο νομάρχης δεν τα καταφέρνετε και εγώ υιοθέτησα διατάξει ώστε να μπορέσει η Γαλλία να υιοθετήσει τα δικά της αυτά που της αντιστοιχούσαν. Για να λάβω μια επιχορήγηση 50% έπρεπε να ξεκινήσω δαπάνες που δεν θα έκανα παλιά. Δηλαδή έρχεται μια στιγμή όπου ο μηχανισμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα η Ευρώπη να δημιουργεί δημόσιες δαπάνες. Παράδοξο. Για ώστε να πάρεις αυτό που σου αντιστοιχεί. Οπότε τελικά να αναρωτιέμαι κατά πόσο υπερβάλλουμε λίγο εδώ, μήπως το παρακάνουμε. Διότι καλό είναι να παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα, αλλά αυτό δεν χρηματοδοτεί στο 100% εκτός ε, ελάχιστες εξαιρέσεις. Και πιστεύω ότι μια τροχοπέδη στην ίσπραξη των όσων μας διαθέτει η Ευρώπη, μπορεί να μας διαθέσει, είναι ότι οι φορείς πρέπει να χρεωθούν για να ανακτήσουν τα κονδύλια. Ίσως λοιπόν κάποια κράτη-μέλη να δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν ε, τα ε, χρήματα που δικαιούνται, διότι κάποια χρονική στιγμή τελικά ε, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν χρηματοδοτεί η Ευρώπη το 100% των δαπανών. Αυτή λοιπόν, ε, η, αυτός ο αγώνας λοιπόν δρόμου εξηγεί τις δυσκολίες που έχουν κάποια κράτη-μέλη να εισπράξουν τα κονδύλια που υπάρχουν στη διάθεσή τους. Και εκεί πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι θα τα αξιοποιήσουμε και θα τα χρησιμοποιούμε όλα. Κάποια χρονική στιγμή υπάρχει κίνδυνος ε, να δημιουργούνται ε, δαπάνες μη αναγκαίες. Ο καθένας κάνει το δικό του, αλλά υποψιάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να γεννά κρατικές δαπάνες. Ενδεχομένως μη αναγκαίες. Τον θα αφήσουμε έτσι αυτή τη φούσκα να δημιουργείται είναι σαν κερδοσκοπία. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να ξεφουσκώσει αυτή η φούσκα και να προσαρμόσουμε κάπως καλύτερα τις πιστώσεις ε, που διαθέτουμε στα κράτη-μέλη. Ε, Ο Ευχαριστώ. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων πρέπει να τηρούνται. Όταν αυτές μετατρέπονται σε πληρωμές, τότε τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι διατεθειμένα να πληρώσουν. Εμένα μου φαίνεται προφανές αυτό. Κάτι άλλο τώρα όταν έχουμε τον κανόνα νησιν 2 ή νησιν 3 Ό,τι και από τα δύο, ό,τι από τα δύο και να έχουμε θα υπάρχουν υπόλοιπα προς εκαθάριση. Γιατί εκπλήσεστε. Υπάρχουν, ε, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν οι ε, υπόλοιπα προς εκαθάριση. Είτε ακολουθούμε τον κανόνα νησιν 2 είτε τον κανόνα νησιν 3 και γνωρίζουμε ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχή ε, Είτε έχουμε τον κανόνα νησιν 2, είτε έχουμε τον κανόνα νησιν 3, δεν θα σταματήσει το 2020, αλλά το 2023. Και ίσως πολλά κράτη-μέλη να γνωρίζουν ότι θα έρθουν ε, ένα σωρό λογαριασμοί το 2020 και το 2021 και που θα πρέπει να πληρωθούν πολλά τιμολόγια και ίσως δεν χρειάζεται να πιεστούν για να συμφωνήσουν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή είναι η λάθος ε, συνέπεια. Όταν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για να πληρώσουμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, προσπαθούμε να καθυστερήσουμε τη δημιουργία νέων προγραμμάτων κτλ. Και μετά τα νέα προγράμματα και η πολιτική συνοχή, η νέα πολιτική συνοχή δεν θα ξεκινήσει το 2021, θα ξεκινήσει το 2023. Και μετά, σε όσου δεν αρέσει η πολιτική συνοχή, αυτοί θα πούν: Κοιτάξτε, κάτι καθυστερήσει, δεν εκτελείται τίποτα και όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Θα μπορούσαμε να επιλύσουμε μια χαρά όλα αυτά τα ζητήματα αν αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευτεί ε, έχουν πληρωθεί και τα κράτη-μέλη όταν δεν πληρώνουν διότι υπάρχει καθυστέρηση εκτέλεσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πληρώσουν και υποχρεούνται να πληρώσουν στο μέλλον για αυτά για τα οποία είχαν δεσμευτεί. Υπάρχει και κάτι άλλο όσον αφορά την ποιότητα των ε, έργων διότι τα κράτη-μέλη επειδή δεν πραγματοποιούν εκτέλεση όπως θα έπρεπε και η εκτέλεση των κρατών μελών σε θέματα ταμείων συνοχής ε, πράγματι δεν είναι καλή, αλλά ω ε, ως επιτοπλίστων ακολουθεί τους κανόνες ε, και ακολουθεί κυρίως τον κανόνα νήσιν 3, σε τελική ανάλυση θα υπάρξει μια πίεση και τελικά κάθε κρατος θα πει ποιο είναι αυτό το έργο που μου τρώει όλα τα λεφτά που ήθελα να δαπανίσω και τελικά εκεί θα έχουμε συνέπεια χειρότερη ποιότητα των έργων, κάτι που πρέπει να αποφύγουμε, γιατί αυτό που επιδιώκουμε είναι η αποτελεσματικότητα ε, και τα καλά αποτελέσματα κάθε έργου. Κυρία Τερτομπλουμ, στον πίνακα στη σελίδα, δεν θυμάμαι ποια σελίδα, ε, με τα ωραία χρώματα. Βλέπουμε την εξέλιξη των ΡΑΛ αναπολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και βλέπουμε αυτό που είναι σε μπλε θα πρέπει να σταματήσει το 2000 και στο 7ο έτος έχουμε μπλε. Ξεκολουθούμε να έχουμε μπλε. Το ίδιο για το 2000-2007. Βλέπουμε το πορτοκαλί να υπερβαίνει το 2014. Και το ίδιο για το 2007-2014. Αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας νήσιν 3 δεν τηρείται. Ναι, έχουμε έργα και από το 1994 που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. 94, ναι. Πρέπει να συνεχίσουμε στα αγγλικά τώρα γιατί η δερμηνία θα σταματήσει. Aurel, from the DG budget, please. Thank you, uh, Mrs. Gressler. And uh, let me start by thanking, first of all, uh, Mevrouw Turtelboom and her team for the good quality of the report and the excellent collaboration uh, with the Commission in the preparation. That was much appreciated uh, on our side. Um,